Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πρακτικά της χθεσινής ε, συνεδρίασης ε, είναι διαθέσιμα. Θέλει κάποιος να σχολιάσει οτιδήποτε επί του θέματος, αν όχι εγκρίνονται τα πρακτικά.